Ja, vielen herzlichen Dank äh, für diese erneute Ansage und ich bedanke. Σας ευχαριστώ πολύ για την νέα αυτή ανακοίνωση και λυπούμαστε ιδιαίτερως που κατέστη για άλλη μια φορά απαραίτητη, λέει η Πρόεδρος. Ιδιαίτερα με τη δουλειά σας. Χωρίς εσάς, χωρίς τους Γερμανείς δεν θα ήταν δυνατή η δουλειά μας εδώ και γι' αυτό εξ ονόματος όλων των συναδέλφων πιστεύω. Μιλώ όταν λέω ότι ελπίζουμε σε μια ικανοποιητική λύση του ζητήματος για όλους τους εργαζομένους. Για να μπορούμε να στηριζόμαστε στην δουλειά σας που είναι απαραίτητη για μας εδώ. Και σας διαβεβαιώ ότι προσπαθούμε πάντα να ολοκληρώνουμε τις συνεδριάσεις μας εγκαίρως και ή δυνατόν και λίγο νωρίτερα και οπωσδήποτε και σήμερα αυτό θα συμβεί. Συνεχίζουμε λοιπόν με το σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης. Έχετε αντιρρήσεις, προτάσεις για τροποποίηση. Αν όχι, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και περνώ στο σημείο 3 έγκριση των πρακτικών της δεκάτης είναι στα, στα έγγραφά σας, δεν βλέπω παρατηρήσεις για τα πρακτικά και προτείνω όπως πάντα να εγκριθούν εάν δεν υπάρχει εκδήλωση αντιρρήσεων με στη διάρκεια της συνεδρίασης. Σημείο 4. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχουμε τις εξής γλώσσες στη Διερμηνία, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ισπανικά, ε, Ελληνικά, Τσεχικά, Πορτογαλικά, Ουγγρικά, Εστονικά, Πολωνικά, Σλοβενικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά. Ε, έχουμε μεταδοση από το διαδίκτυο όπως πάντα και θέλω να σας υπενθυμίσω την διάσκεψη υψηλού επίπεδου της 26ης Ιουνίου για την πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος Ταγιάννη σε συνεργασία με την Επιτροπή μας ε, έχει αναλάβει ε, υπό την αιγίδα του αυτή τη συνεδρία σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, πολιτιστική κληρονομιά, από τις 2 μέχρι τις 7 το βράδυ στην αίθουσα της Ολομέλειας και με παρουσία του Πρόεδρου Γιουνκέρ, ε, Υπουργών Αρμόδιων για θέματα πολιτισμού, επιφανών προσωπικότητων και εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα πολιτισμού. Έχετε το πρόγραμμα. Σας το έχουμε στείλει με το ε, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υπάρχει και ο σχετικός σύνδεσμος για να ε, δηλώσετε έως τις 19 του μηνός ε, την συμμετοχή σας. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω πως στις συνεδρίες των συντονιστών ενημέρωσα τους συντονιστές, τους συναδέλφους, ότι λόγω της ε, περιορισμένης μερικές φορές ε, παρουσίας συναδέλφων σε εκδηλώσεις της Επιτροπής μας και κυρίως όταν έχουμε εδώ προσκεκλημένους, έχω αναλάβει την πρωτοβουλία να αναλάβω πιο σκληρά μέτρα και έτσι να περιορίσω τις εργασίες της Επιτροπής μας στη νομοθετική δουλειά και ε, ακροάσεις θα διεξάγονται μόνο όταν οι συντονιστές με ενημερώνουν και με διαβεβαιώνουν προκαταβολικά ότι θα είναι επαρκής η παρουσία των συναδέλφων των οποίων τα ονόματα θέλω να μου, να μου κοινοποιούνται προκαταβολικά. Παρακαλώ λοιπόν ήδη αυτήν την εβδομάδα να μας αποστείλετε μια, ε, ένα μήνυμα ηλεκτρονικό για να ξέρουμε ποιοι θα είναι οι ε, βουλευτές που θα λάβουν μέρος σε μια ακρόαση προγραμματισμένη για τις 11 Ιουλίου. Εάν τυχόν και δεν είναι επαρκή ο αριθμό των παρόντων, με λύπη μου θα χρειαστεί να την ματαιώσω, διότι βρίσκω πολύ δυσάρεστο να έχουμε εδώ προσκεκλημένου και να μην έχουμε αρκετούς βουλευτές. 31 είναι οι βουλευτές τακτικά μέλη, άλλοι 31 οι αναπληρωτέ. Ε, καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος ε, να λείπει για κάποιο λόγο, αλλά δεν μπορεί να εκπροσωπεί 31 τακτικά μέλη ένας βουλευτής. Γι' αυτό είμαι αναγκασμένη να προβώ σε πιο δραστικά μέτρα. Επίσης, για τους εισηγητές που εξετάσαμε μάλιστα σε σχέση με τα προγράμματα την προηγούμενη εβδομάδα και δείτε προγράμματα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής αλλά και κάθε γνωμοδότηση, όχι μόνο δηλαδή τις εκθέσεις μας. Παρακαλώ λοιπόν να επαληθευτεί αυτό για να ξεκινήσουμε το χέτερο δυνατό τη δουλειά μας. Δεν έχουν λυθεί όλες οι συγκρούσεις αρμοδιοτήτων αλλά πιστεύω παρόλα αυτά ότι όποιος μπορεί, όποιος είναι εισηγητής και μπορεί ήδη να ξεκινήσει τη δουλειά του, να ε, ετοιμάσει να ε, διατυπώσει κάποιες σκέψεις για το τι, ποιο θα είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλει να αποστείλει με την έκθεσή του και συνολικά αν θέλετε οι αρμόδιοι εισηγητές για όλες τις εκθέσεις να μπορούμε να ε, ξέρουμε τι είναι να κατατεθεί για έγκριση στην Επιτροπή μας. Ας ξεκινήσει λοιπόν αυτή η δουλειά το ταχύτερο δυνατό για να μην χάσουμε τον έλεγχο του χρονοδιαγράμματός μας. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις μου. Και τώρα, με χαρά, καλώς ορίζω τον Επίτροπο Ναύρατσιτς, ο οποίος θα έρθει να, ήρθε για να μας ε, παρουσιάσει τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, ένταξη του πολιτισμού στο επίκεντρο των ε, δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια θα μας εκθέσει και το γενικότερο υπόβραβαθρο, που αφορά τις δύσκολες διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μάλιστα ένα χρόνο πριν από τις προσεχείς ευρωεκλογές. Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει προσπάθειες για ένα ε, πλαίσιο για την εκπαίδευση στο 2025, αλλά και για τον πολιτισμό, για τη συμμετοχή των νέων και την υποστήριξή τους στα πολιτιστικά αγαθά, στρατηγική για τους νέους, ε, θεματολόγιο για τον πολιτισμό. Είναι όλα αυτά τα θέματα τα οποία προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε και νέες προτάσεις προγραμμάτων για το προσεχές δημοσιονομικό, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, για τον ε, για το δε πρόγραμμα Εράσμου, βλέπουμε διπλασιασμό του προπολογισμού του με ικανοποίηση. Είδα σήμερα νωρίτερα εκπροσώπους της γερμανική κυβέρνηση, του οποίους και εξέφρασα την ικανοποίησή του μου, την ικανοποίησή μου γιατί είναι η πολύ ικανοποιητική η ανακοίνωση από πλευρά του κυρίου Γιουνκέρ, του Προέδρου, στην ε, ομιλία για την κατάσταση της Ένωση για πολλαπλασιασμό, εννέα πλασιασμό συγκεκριμένα των ποσών για τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε να κάνουμε πλέον με 26 εκατομμύρια, με πιο συγκεκριμένε προτάσει, που βέβαια δεν ήταν αυτό το οποίο θέλαμε, αυτό που περιμέναμε, αυτό που έχει ζητήσει βέβαια το Κοινοβούλιο με το ψηφισμά του, μεν... Και γι' αυτό θα χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε Πάντως, σε αυτή την ε, συζήτηση σήμερα με σας κύριε Επίτροπε, θα ήταν καλό να περιοριστούμε στα εγκάρσια ζητήματα. Για το Εράσμους και το πρόγραμμα για τον πολιτισμό αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ίσως μπορούμε να πούμε περισσότερο στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα η σημερινή μας συζήτηση ιδιαίτερα να δώσει έμφαση στα πιο γενικά και εγκάρσια ζητήματα. Έχω επανειλημμένω επισημάνει την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει τον ακτήριο λακτισμα για, την, ε, για τον χώρο πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι Υπουργό Μεταφορών ε, για την εκπαίδευση, συγγνώμη, και μάλιστα πρέπει να σα πω ότι Υπουργό Μεταφορών τη Γερμανία, εκπρόσωπο Υπουργείου Μεταφορών τη Γερμανία ε, από τοπικό κρατήδιο, με ρώτησαν πρέπει να φοβούνται οι Γερμανοί που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδιότητε ή πρωτοβουλίε για την εκπαίδευση. Εγώ ε, γέλασα βέβαια, αλλά του είπα ότι ίσω τελικά δεν είναι κακό να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εκπαίδευση και μέσα σε αυτό ίσω μπορέσουν τα κράτη-μέλη να δεσμευθούν αμοιβή βέβαια ε, να ε, τηρείται βέβαια πάντα η αρχή της επικουρικότητας, αλλά ταυτόχρονα και να προχωρήσουν από κοινού. Και έτσι τα κρατη αλλά και τα κρατήδια της Γερμανίας ε, δεν είναι ανάγκη πάντα να ξεσηκώνονται λέγοντας όχι μακριά τα χέρια από την εκπαίδευση. Ίσως μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάποια πρόοδο στον χώρο αυτόν και γι' αυτό καταρχάς σας ευχαριστώ για την ε, πρώτη αυτή πρόταση και δεύτερον σας δίνω το λόγο για να μας δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως είπα, εγκάρσια για το χώρο της εκπαίδευσης, για, την, ε, για τον πολιτισμό, την νεολαία, τον προγραμματισμό σας και τις κατευθύνσεις όπως τη σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ναύρατσιτ, χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε εδώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τον περασμένο Νοέμβρη ε, έγινε η τελευταία συνάντηση του διαλόγου και είχα πει ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να θέσει καινούριου φιλόδοξους στόχους για τον, τους τομείς Σήμερα μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι πράγματι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός βρίσκονται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντα. Ε, υπάρχει μια ομοσυνένεση πλέον ότι έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο για να δημορφωθούν δίκες και ισότιμες κοινωνίες. Έχουμε την όρμη, πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Στο τέλος ε, του περασμένου χρόνου στείλαμε ένα... Ε, το, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από εμά μια πιο ενισχυμένη προσπάθεια και προσπαθούμε να θέσουμε αυτέ τι πολιτικέ στο κέντρο των προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι τα καταφέραμε και ευχαριστώ πολύ για την στήριξή σα. Πώ προωθεί αυτή την εντολή η Κομισιόν. Την περασμένη Νοέμβρη εκδώσαμε ε, μια ανακοίνωση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Ε, την δεχτήκατε πολύ θετικά εσείς. Από τότε και μέσα σε έξι μόνον μήνες ε, υποβάλαμε προτάσεις για ε, διάφορα θέματα ε, του 2025 για τη δημιουργία ενό, μιας, ε, ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης που θα πρέπει να στηρίζεται σε τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, ε, μια προσέγγιση διαβίου μάθησης και μια ευρώ, ευρύτερη έννοια της εκπαίδευσης για όλους. Όπως το είπατε και εσείς στο ψήφισμά σας για τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, η, μάθηση ξεκινάει νωρίς και συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Δεύτερον, ισχυρά θεμέλια. Οι έρευνες δείχνουν ότι το 20% των 15 χρονών αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να διαβάσουν, να γράψουν ή να χειριστούν τα βασικά μαθηματικά σωστά. Ε, αυτό έχει σχέση με τον κοινωνικό εξοπλισμό, αλλά όχι μόνο. Οι νέοι ε, αυτοί οι νέοι δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα που θα τους κάνουν ανταγωνιστικούς σε μια ανταγωνιστική Ευρώπη. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι μας θα έχουν τις βασικές δεξιότητες για να χτίσουν το μέλλον τους. Και τα ισχυρά θεμέλια επίσης έχουν σχέση και με τις ε, κατάλληλες αξίες και συμπεριφορές. Τρίτο στοιχείο είναι η δεκτικότητα. Θέλουμε μια Ευρώπη όπου οι νέοι μας ε, θα έχουν ως κανόνα το να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να δουλέψουν, να μάθουν, να κάνουν εθελοντισμό κλπ. Μόνο έτσι θα χτίσουμε μια πραγματικά ισχυρή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Για να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά, αρχίσαμε να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρώτη, για την οποία είμαι ιδιαίτερα περήφανο ε, είναι μια σύσταση προ τα κράτη-μέλη για τις κοινέ αρχές, ε, την εκπαίδευση για όλους και την ευρωπαϊκή διάσταση της ε, δασκαλία. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι θα μαθαίνουν ο ένα για τον άλλον και για τον εαυτό τους, έτσι ώστε όλοι να κινούμαστε προ την ίδια κατεύθυνση και θέλουμε επίσης να μαθαίνουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το λαϊκισμό, το διχ, τις προσπάθειες διχασμού ε, και την παραπληροφόρηση. Χαίρομαι που οι Υπουργοί την έκαναν δεχτεί αυτή τη σύσταση. Ποτέ στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε καταστήσει τόσο σαφές πόσο σημαντική είναι η προώθηση των κοινών μας αρχών προκειμένου όλοι να ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να νιώθουμε ότι ανήκουμε και να μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές από οπουδήποτε και αν προερχόμαστε κοινωνικά. Ο ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευση σημαίνει ότι όλοι θα έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες έτσι ώστε να πετυχαίνουν το σκοπό του. Γι' αυτό το λόγο πρότεινα ε, μια ε, καινούργια σύσταση για τις ε, βασικέ δεξιότητε. Ε, τεχνολογία, ε, μηχανική, μαθηματικά ε, και επιστήμες. Και χαίρομαι που και αυτή η σύσταση ήδη οθετήθηκε από τα κράτη-μέλη. Επίσης υπέβαλα ένα πρόγραμμα ψηφιακής δράσης με, με τρεις στόχους. Να στηριχθεί η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της εκπαίδευσης για μέσω καλύτερης ανάλυσης των δεδομένων και πρόβλεψης. Το στηρίζουμε με το online εργαλείο Selfie που θα επιτρέπει στους φοιτητές, στους μαθητές και τους δασκάλους και καθηγητές να υποφεληθούν της τεχνολογίας. Κατόπιν υπέβαλε και ένα δεύτερο πακέτο τον περασμένο μήνα με τρεις συστάσεις συμβουλίου μια καινούργια στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την νεότητα, μια νέα ατζέντα για τον πολιτισμό και μια ανακοίνωση για την ενίσχυση τη Ευρώπη. Ε, το χτίσιμο μια πιο ενισχυμένη δυνατή Ευρώπη. Βασιζόμαστε στο γεγονό ότι τα πρώτα χρόνια στη ζωή ενό ανθρώπου είναι τα πιο κρίσιμα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει εξ αρχή να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Μόνο έτσι θα βοηθήσουμε την ισότητα και την κοινωνική κινητικότητα. Επίση, υπέβαλα ένα, μια σύσταση για να βελτιωθεί η διδασκαλία και η εκμάθηση γλωσσών. Ο τελικό μα στόχο είναι όλοι να μπορούν να μιλούν τουλάχιστον δύο γλώσσες πέραν της μητρικής τους στο τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Οι γλώσσε ανοίγουν πόρτες, μα επιτρέπουν να βρούμε απασχόληση και μας επιτρέπουν επίση να αλληλοκατανοούμαστε. Είναι το κλειδί για να ανακαλύψουμε την πυκλομορφία της Ευρώπης και είναι πολύ σημαντικές στο να επιτρέψουν στους νέους να είναι πραγματικά κινητικοί να, ε, και ε, προετοιμασμένοι. Ε, στο ίδιο πνεύμα, το ψήφισμα για την ε, αυτόματη εμβέα αναγνώριση επιτρέπει στους φοιτητές να κινούνται στον, ε, στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Θα επιτρέψει επίσης να ενισχυθεί συνεργασία ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ως τμήμα του ίδιου πακέτου, υπογραμμίζουμε και άλλα βήματα για τη δημιουργία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και της Ευρωπαϊκής ε, Φοιτητικής Κάρτας. Ο νέος ευρωπαϊκός χώρος θα πρέπει πραγματικά να διαθέτει ε, ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με ισχυρά δίκτυα ε, ακαδημαϊκών ε, πανεπιστημιακών ε, ε, ιδρυμάτων που θα εξυπηρετούν την κοινωνία και θα προωθούν την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε την αριστεία στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό βοηθάει και τι οικονομικέ και κοινωνικέ εξελίξει στις περιοχές στι οποίε είναι εγκατεστημένα και προχωράμε με την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής φοιτητικής κάρτας με στόχο να καταστεί πιο εύκολο για τους φοιτητές να ε, κινούνται στο εξωτερικό ε, και, να και να μειωθούν τα διοικητικά βάρη. Αυτά όλα συνδέονται με τα σχέδιά μας για την ενίσχυση της συνεργασίας των πολιτισμών και την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων. Με την νέα μας πρόταση για την νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κουλτούρα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ισχύ του πολιτισμού για την ε, οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε επίσης και στις εξωτερικές μας σχέσεις έτσι ώστε να δημιουργήσουμε πιο ισχυρούς συνδέσμους με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο. Η ευρωπαϊκή, ε, το ευρωπαϊκό έτος πολιτικής κληρονομιάς στην Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει καταλήτη συγγνώμη, 2.560 εκδηλώσει έχουν ήδη οργανωθεί στα κράτη-μέλη με ένα εκατομμύριο συμμετέχοντες και ακόμα έχουμε πολλά που θα οργανωθούν στο μέλλον. Αυτό το έτος ε, ταυτόχρονα θα μας δώσει και την ευκαιρία να εξασφαλίσουμε ότι ο πολιτισμός θα εξακολουθήσει να χαίρει της αναγνώρισης που αξίζει και ότι θα χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία της μελλοντική Ευρώπης. Η Το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική κληρονομιά που θα παρουσιάσει το τέλος του έτους θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διοργανώσατε μια εκδήλωση υψηλού επίπεδου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κληρονομιά στην... στο... που οργανώνεται την επόμενη εβδομάδα στις θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να συζητήσουμε το πώς θα εκμεταλλευτούμε τον υπόλοιπο χρόνο. Θα πρέπει να φτάσουμε κοντά στους ε, νέους μας κατά αυτού του έτους και είναι προτεραιότητα γιατί έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ε, δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας του, ε, του, στο μέλλον. Θα πρέπει όμως να είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό και να τους δοθεί η ευκαιρία να διαμορφώσουν τη δική τους ζωή και τις κοινότητες στις οποίες ζουν. Ε, η ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Στατική Νεότητα που προτείνουμε επίση θα μα επιτρέψει ακριβώς αυτό να πετύχουμε. Πρόκειται για ένα πολύ πιεστικό και επίκαιρο θέμα εξαιτία των επικίνδυνων ευρωπαϊκών εκλογών. Το ε, να συνδέσουμε τους νέους μέσω ε, διασυνοριακών δραστηριοτήτων ελεγγύης ε, τους επιτρέπει να νιώθουν πιο Ευρωπαίοι. Γι' αυτό το λόγο χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για την νομική βάση ε, του ε, Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελον, ε, Αλληλεγγύης και Εθελοντών. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τρόπερ και τους συνεισηγητές ε, που το βοήθησαν. Ε, ως αποτέλεσμα της δικής σας ευελιξίας θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις σύντομα και την Τετάρτη να επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο αυτή η συμφωνία. Ε, η νομική αυτή βάση επιτρέπει περισσότερη χρηματοδότηση και μεγαλύτερες ευκαιρίες ε, στην περίοδο 2018-2020. Όλοι μαζί μπορούμε να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια, αλλά, αυτό χρειαζόμαστε, ε, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε επαρκή χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ό,τι σαν αναλογούσε. Για την περίοδο μετά το 2020 προτείναμε πάνω από, ε, πάνω από διπλασιασμό του προπολογισμού του Εράσμου έτσι ώστε να αποφελθούν πάνω από δύο φορές ε, ε, ο αριθμός των νέων που ε, σήμερα. Ε, έχουμε επίσης προ, αύξηση του προπολογισμού του, της Ευρώπη Ευρώπης κατά 25%. Σε άλλα προγράμματα βέβαια έχουμε μειώσεις και ε, μικρότερες αυξήσεις. Ε, ε, εδώ όμως προσπαθούμε ε, να επιτύχουμε μια εξέλιξη, όχι μια επανάσταση. Θέλουμε τα προγράμματά μας να φτάνουν σε περισσότερους ανθρώπους, για παράδειγμα στους μειονεκτούντες πληθυσμούς, καθώς επίσης και να δώσουμε σε μαθητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Θέλουμε να ανοίξουμε τα προγράμματά μας σε μικρότερες οργανώσεις, με μικρότερες πιο στενές εταιρικέ σχέσεις και πιο απλοποιημένες διαδικασίες. Θέλουμε το μελλοντικό πρόγραμμα Εράσμους να γίνει πιο διεθνές, με περισσότερες ευκαιρίες ε, σε μαθητές ε, σε φοιτητές ε, να αποκτήσουν εμπειρίες και εκτός Ευρώπης. Επίσης θα ενισχύσουμε την κινητικότητα στον αθλητισμό και θα ενισχύσουμε την στήριξή μας σε σχέδια τα οποία θα μας επιτρέψουν ε, να ε, προστατέψουμε το, ε, τον, τον αθλητισμό. Επίσης θα διευκολύνουμε τις συνέργειες μεταξύ του Εράσμους και άλλων προγραμμάτων όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πρόγραμμα ΣΥΝ. Ξέρω ότι ανησυχείτε για το θέμα του στο τόπο του Εράσμου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Έτοιμο. Για να δημιουργήσουμε την Ευρώπη, οι κοινοτομίε είναι βασικό για τους ε, καλλιτέχνες, τη μουσική, τους καλλιτέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά. Ε, στα ΜΜΕ, περισσότερα χρήματα επενδύονται για τη διεθνή προώθηση και διανομή των ευρωπαϊκών έργων και καινοτόμων ε, αφηγημάτων μαζί με τις ευρωπαϊκές, ε, θα δημιουργηθούν ευρωπαϊκές εταιρείες για να ενισχύσουμε την ορατότητα της ε, ευρωπαϊκής προσπάθειας. Ε, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά το 2020 θα λάβει υπόψη την, τα, αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για την τρέχουσα πρόταση. Επιπλέον, θέλω να συμπεριλάβω το, το πρόγραμμα για τους Ευρωπαίους εθελοντές. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ε, θα συγκεράσει όλες τις ευκαιρίες που προσφέρουμε σε νέους ανθρώπους για να προωθήσουν δραστηριότητες αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Για να ολοκληρώσω. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε σαφείς ε, τολμηρούς στόχους και έναν προπολογισμό που μας δίνει τα μέσα για να το υλοποιήσουμε όλο αυτό. Πιστεύω ότι οι προτάσεις που ε, παρουσίασα είναι καλή αφετήρια. Είμαστε στην αρχή μιας θαυμάσιας νέας εποχής. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Πρέπει να αναπτύσσουμε τις ιδέες μας, ειδικά για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ας πούμε. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι δεσμεύσεις που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη μεταφράζονται σε απτά ωφέλη για τους πολίτες. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης ότι ο ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης δεν είναι ένα μακρινό όραμα, αλλά γίνεται πραγματικότητα. Και μαζί θα πρέπει να στηρίξουμε τις προτάσεις για τα, προγραμματά, για τα προγράμματά μας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είμαι σίγουρος ότι θα έχω την υποστήριξή σας. Ε, περιμένω να ακούσω τώρα τις απόψεις και να τις συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο Ναύρατσιτς. Και τώρα παρακαλώ τους συντονιστές να λάβουν το λόγο. Το πολύ για τρία λεπτά ο καθένας. Με τη διαδικασία ping-pong, την ξέρουμε καλά πια. Ερώτηση ή τοποθέτηση και απάντηση. Ακούμε πρώτα τους συντονιστές και μετά τους λοιπούς συναδέλφους. Κύριο Στρογεύσκη πρώτος λοιπόν. Έχετε το λόγο. Τρία λεπτά το πολύ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με τα καλά νέα. Το Erasmus Plus, πάνω απ' όλα. Είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα με, τη μεγαλύτερη έγκλη και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά και τους πόρους που έχει. Και χαιρόμαστε που στις επόμενες, στο επόμενο πουδουμού, πουδουπού θα υπάρξει διπλασιασμός του προϋπολογισμού του και όλες οι γλώσσες θα έχουν συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αυτό το πρόγραμμα και δεν θα πρέπει να δίνουμε προτίμηση στις κλασικές γραμμές προπολογισμού, αλλά στις ολοκληρωμένες. Κάτι που είναι σημαντικό και το τονίζουμε συχνά είναι ότι όλες οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται με αποτελεσματικό τρόπο στον τομέα μας συχνά συσσωρεύουμε καθυστερήσεις στον χώρο τη εκπαίδευση. Σήμερα οι δικαιούχοι οι οποίοι παραπονούνται για καθυστερήσεις βέβαια είναι λιγότεροι. Ε, υπάρχει μια βελτίωση. Σε ό,τι αφορά για την Ευρώπη, για τους πολίτες και την δημιουργική Ευρώπη, υποστηρίζουμε ότι ένα ποσοστό χαμηλό λαμβάνει μια συγχρηματοδότηση 11-12%. Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί δικαιούχοι που δεν ικανοποιούνται. Επομένως, τα προγράμματα πρέπει να βελτιωθούν και βελτιώνονται, αλλά πολύ πολύ αργά. Σε ό,τι αφορά το μήνυμά σας ή τα μηνύματά σας γενικά, Επίτροπε, πιστεύουμε ότι πολλά σημεία είναι ικανοποιητικά και αυτό μας ευχαριστεί. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Thank you. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Ο βασικός μας στόχος και η στόχη πολιτικής για την επόμενη περίοδο, για το επόμενο πουδουπού, είναι το Εράσμος να είναι πιο προσπερλάσιμο από όλους. Να έχει μεγαλύτερη κοινωνική έλξη και έγκλη και να είναι πιο προσβάσιμο σε κοινωνικά μειονεκτούντες ανθρώπους. Γεωγραφικός πώς ξέρουμε ότι το Εράσμος σε μερικές χώρες προορίζεται για τις ε, μεσές ή, και ανώτατες τάξεις. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να διευρύνουμε την κοινωνική βάση, να είναι πιο προσπελάσιμο από περισσότερους ανθρώπους και άλλων εισοδηματικών και κοινωνικών τάξεων και ακριβώς γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μεταφράσουμε όλες ε, τις σχετικές πληροφορίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Γιατί μερικές φορές τα βάρη δεν είναι μόνο υλικά αλλά και άλλα. Θέματα γλώσσας ε, και άλλες δυσκολίες. Η Δημιουργική Ευρώπη μαζί με τον ορίζοντα 2020 ήταν από τα πιο ελκυστικά προγράμματα με πάρα πολλούς ε, συμμετέχοντες, ε, ετούντες κτλ. Η μικρή αύξηση του προϋπολογισμού δεν πρόκειται να λύσει όλα τα προβλήματα όμως, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προστατεύσουμε, να παραμείνει αυτόνομο πρόγραμμα. Έχουμε μια δυνατότητα για ένα χωριστό πολιτιστικό πρόγραμμα. Φυσικά δεν είναι απομονωμένο, γιατί θα πρέπει να συνδέεται με άλλα προγράμματα προφανώς και να τους κρατήσουμε αυτούς τους δεσμούς. Με το πρόγραμμα χειραφέτησης, με το πρόγραμμα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων κτλ. κτλ. Αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε μία αυτόνομη χρηματοδότηση για τα πολιτιστικά προγράμματα. Για το πολιτιστικό πρόγραμμα. Στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού το πιο σημαντικό θέμα του Creative, ε, Creative Europe είναι η κινητικότητα των καλλιτεχνών. Χρηματοδοτούμε προγράμματα κινητικότητας των καλλιτεχνών και θα το κάνουμε και στο μέλλον και πιστεύουμε ότι η αύξηση αυτή του προϋπολογισμού θα είναι πιο ικανοποιητική και για σας και για τα κράτη-μέλη και τους ΜΚΟ και για τις διάφορες ενδιαφερόμενες κοινότητες. Ευχαριστώ. Κυρία Κώστα, μία πολιτική γενική κρίση που μου φαίνεται σημαντική. Στη δεύτερη Το δεύτερο τμήμα της νομοθετικής περίοδου, τα δυόμιση χρόνια αυτά, είδαμε μια νέα φάση να δημιουργείται. Δηλαδή, οι πολιτικές για την ευρωπαϊκό χώρο ε, εκπαίδευσης, που σημαίνει σύγκληση δεν σημαίνει ταύτιση, μέσω ε, ίσων ευκαιριών, κινητικότητας, κοινών αξιών κτλ. Ε, τονώθηκαν, προωθήθηκαν. Αυτό αναγνωρίζεται, αλλά και έγινε και χάρη στη δουλειά που έκανε το Κοινοβούλιο. Από την άλλη, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Δημιουργική Ευρώπη, εκεί θα δούμε κάποια πιο σημαντικά πράγματα. Οι ψηφιακέ ικανότητε, η, συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Connect, ε, μας δίνει πολύ πιο απτούς στόχους αυτή η συνεργασία. Τα προγράμματα σήμερα είναι εργαλεία μαζί με το θεματολόγιο και το θεματολόγιο για τον πολιτισμό, αλλά και τα προγράμματα, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνάφεια ε, για να υλοποιούμε αυτούς τους στόχους. Αυτό είναι το γενικό. Βέβαια υπάρχει και το θέμα του προπολογισμού, πάντα ανεπαρκή είναι. Αυτή η πολιτική λοιπόν θα πρέπει να μπει στο κέντρο τη προσπάθεια. Το Κοινοβούλιο σα έχει δώσει πάρα πολλέ ενδείξει και σα έχει υποστηρίξει. Τώρα, δύο ερωτήσει για το ένα πρόγραμμα και δύο για το άλλο. Ε, για το Erasmus Plus, ξέρουμε ότι στα χαρτιά υπάρχουν 26 δισεκατομμύρια, όχι 30. Αλλά πέρα από αυτό τα πράγματα είναι θετικά. Εμείς ε, επιμένουμε για την αύξηση των κονδυλίων. Υπάρχουν όμως και, συ, και γραμμές οι οποίες ε, αφορούν το Discovery You. Ε, καθώς και νέες σημαντικές ε, δράσεις για την κινητικότητα στα, στην ανώτατη εκπαίδευση και στα δίκτυα των πανεπιστημίων. Τώρα, ε, για την εκπαίδευση των ε, ενηλίκων. Υπάρχει μεγαλύτερη επικέντρωση. Το Erasmus Plus θα θέλαμε να, ε, θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη αυτονομία. Το είχαμε ζητήσει από πριν. Τώρα, για, το, για την κάρτα για τους φοιτητές. υπάρχουν ε, κάποιες διευκολύνσεις. και το Creative Europe, δύο ερωτήσεις. Αύριο θα συζητήσουμε τα προγράμματα βέβαια, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω τώρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι θετικό το γεγονό ότι πολλέ από τι ενδείξει του Κοινοβουλίου τις έχετε λάβει υπόψη και του εισηγητή και γενικά όλων. Ε, Παραδείγματο χάρη την κινητικότητα των καλλιτεχνών, ε, ε, μουσική, πολιτιστική κληρονομιά, ε, σχέδιο, μόδα κτλ. Όλα αυτά πολύ σημαντικά. Είναι φιλόδοξε οι προσπάθειές σα, μα ενδιαφέρουν, Όμω οι πόροι δεν είναι Α κάνουμε μια περισσότερη προσπάθεια σε επίπεδο πόρων. Διερωτώ λοιπόν, και εδώ είναι το ερώτημα, γιατί επιλέξατε να μην, να μην τα ονομάζετε προγράμματα, αλλά strand. Ε, όταν έχουμε ένα πρόγραμμα, τα πράγματα είναι πολύ πιο διαρθρωμένα. Και δεύτερον, δεν μας ε, η επιλογή για τις ποσοστώσεις του προπολογισμού. Γιατί λέει πάντα μέχρι το τάδε, ας πούμε, ποσό. Δεν είναι σωστό. Γιατί μπορεί αυτό το μέχρι το μπορεί να είναι πολύ λίγο. Καλό θα ήταν να μας δώσετε ποσοστά. Μαζί με το μέχρι το συγκεκριμένο ποσό, ας πούμε. Ή μάλλον, διορθώνει ομιλήτρια, όχι λιγότερο από και τις ποσοστώσεις. Αλλιώς δεν ξέρουμε πώς κατανέμονται οι πόροι ανάμεσα στους τρεις τομείς. Επίτροπος. γνωρίζω τις υποχρεώσεις μου όπως προλέγονται από τις συνθήκες και ξέρω ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνω στην εκπαιδευτική ή την πολιτιστική πολιτική των κρατών μελών. Όμως, ταυτόχρονα μπορώ να ε, ξεκινώ δράσεις οι οποίες προσθέτουν ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Κατά την άποψή μου όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν προστιθέμενη αξία, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στον τομέα τη εκπαίδευση, αλλά και στον τομέα του πολιτισμού. Και ποια είναι αυτή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Είναι αυτή που ε, προκύπτει ως πρόσθετη εναντί του αθρίσματος των προσπαθειών των κρατών μελών. Ε, έχουμε κάποιους κοινούς στόχους, αυτούς εντοπίζουμε και προτείνουμε συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Νομίζω ότι ο ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης μπορεί να είναι το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής εκπαίδευσης με πλήρη σεβασμό βέβαια της ανεξαρτησίας και αυτονομίας των κρατών μελών. Στον εντοπισμό συγκεκριμένων στόχων και συγκεκριμένων δράσεων. Επί του παρόντος, ε, οι αντιδράσεις των κρατών μελών ήταν πολύ θετικές και στο project και στο σχέδιο για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ε, και στο σχέδιο για τον ενιαίο εκπαιδευτικό χώρο στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία αυτής της συνεργασίας. Το ίδιο και στη χρηματοδότηση. Το έρασμος είναι το, αυτό που περισσότερο γνωρίζουμε. Ε, αλλά δεν είναι το μόνο που αυξάνει τον προπολογισμό του και η Δημιουργική Ευρώπη και ο Ρίζοντας 2020 αυξάνει τον προπολογισμό τους. Και σίγουρα μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα αν χρησιμοποιήσουμε παρόμοιες ε, πρωτοβουλίε άλλων προγραμμάτων, για παράδειγμα για τα πανεπιστήμια. Ο Ορίζον 2020, ο Ορίζον Ευρώπη στο μέλλον, ε, έχει παρόμοια προγράμματα τα οποία, μπορούν να, τα οποία μπορούμε να αποφεληθούμε ή στην πολιτιστική πολιτική, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, έχει δραστηριότητες και σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και ε, ορισμένα προγράμματα επιχειρηματικότητας στον αθλητισμό, στη, στις, ε, στην απόξη δεξιοτήτων αθλητισμού. Οπότε μπορούμε και αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε για χρηματοδότηση. Το ίδιο ισχύει για την Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα. Θα χρηματοδοτηθεί εν μέρη από το έρασμος, αλλά και από την διευκόλυνση συνέδοντας στην Ευρώπη, που ε, έχει ως στόχο την κινητικότητα. Συνδέοντας αυτά τα δύο μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ κύριε Μπίλτ. Παρακαλώ. Ε, ζητώ συγγνώμη δεν έβρισκα το κουμπί μου. Ε, πρόεδρε ευχαριστώ. Κύριε Ναύρατσος, ευχαριστώ για τις εξηγήσεις. Ο Γύρκη Κάτενεν, αντιπρόεδρος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε ότι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρώπης ήταν το ότι έχτισε γέφυρες ανά την Ήπειρο με τη δημιουργία ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων και των πολιτών. Ωστόσο, παρα, παρεμποδίζουν ακόμα την κινητικότητα στην εκπαίδευση πολλά εμπόδια Δυστυχώ η κινητικότητα που επιδιώκεται με έναν ευρωπαϊκό χώρο για την εκπαίδευση, άλλο στόχο δεν έχει παρά να ετοιμάσει τους εργαζομένους στο να εργάζονται σε χώρα άλλη από τη χώρα προελεύσεω. δηλαδή να είναι όλο και πιο εύπλαστη αυτή και χειραγώγημη. Δεν ικανοποιείται κανένα άλλου τα συμφέροντα παρά μόνο των πολυεθνικών. Όταν ε, αρχίσουν να μετατοπίζουν τις, ε, τις εγκαταστάσεις από τη μία χώρα στην άλλη και βέβαια είναι υποχρεωμένοι οι εργαζόμενοι να το δεχθούν αυτό και με χαμηλότερες αμοιβέ, γιατί οι μετατοπίσεις ε, επιχειρήσεων δεν είναι μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κάνετε τότε το 2011 51% των γαλλικών επιχειρήσεων που ε, μετεγκατέστησαν ε, τις ε, δραστηριότητές τους πήγαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Όλο και περισσότερο ανταγωνισμό δηλαδή προξενείται και οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα πρέπει να εργάζονται πλέον για να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας στους νέους της χώρας προελεύσεως. Έχετε στόχο 40% πτυχιούχους από την εκπαίδευση για το 2020. Για τα αποτελέσματα αυτά όμως θα πρέπει να μειώνεται όλο και περισσότερο το επίπεδο των πανεπιστημιακών πτυχίων και απαιτήσεων. Πιο πολλοί πτυχιούχοι λοιπόν, αλλά με όλο και χαμηλότερης ποιότητας πτυχία. Αποτέλεσμα. Για να έχει κανεί μια ευκαιρία να επιβιώσει στην αγορά εργασία, θα πρέπει να λαμβάνει περισσότερα πτυχία, δηλαδή υπερβολική ε, πρόσβαση, ε, υπερβολικά μεγάλο αριθμό πτυχίων που όμως δεν σημαίνει ότι θα έχουν αυτά αξία. Αντιθέτως θα έχουν όλο και χαμηλότερη αξία. Εξού και η πρόταση για την ε, τεχνική εκμάθηση, για την πρακτική εκμάθηση που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως στόχο με 25% για το 2025. Αυτό δεν αποδεικνύεται. Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο. Όλο και περισσότερη εκπαίδευση λοιπόν με όλο και λιγότερη αξία. Και άρα χρειάζεται και πάλι όλο και περισσότερη εκπαίδευση. Με αυτούς τους στόχους μόνο επιδεινώνονται οι ανισότητες γιατί οι πιο εύποροι μόνο μπορούν να έχουν την πολυτέλεια μακροχρόνιων σπουδών, όπως στη νομική. Δύο μάστερ στη Γαλλία πλέον θεωρούνται δεδομένο, εάν κανείς δεν πάει στα αγγλοσαξονικά κράτη, που χρειάζεται να πληρώνει και 50.000 ευρώ το χρόνο για ένα μάστερ. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ε, κύριε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος όσο η κυρία Βουλευτής. Γιατί βλέπουμε μείωση στην απασχόληση των νέων. Και αυτό οφείλεται σε έναν βαθμό τουλάχιστον και στην οικονομική ανάπτυξη, ακόμη και σε χώρες της Νότιας Ευρώπης. αλλά και σε ένα πιο πρακτικά εφικτό σύστημα εκπαίδευση ορισμένα κράτη. Δηλαδή τώρα κίνητρα για μια εκπαίδευση που εξασφαλίζει δεξιότητε με τον προσανατολισμό τα Μεταρρυθμίσεις σε ορισμένα κράτη προ την κατεύθυνση αυτή έχουν φέρει αποτελέσματα και έτσι βλέπουμε στην επαγγελματική κατάρτιση με το διαδικό σύστημα που έχουν ορισμένε χώρες καλύτερα αποτελέσματα ή επιχειρηματικές ε, δραστηριότητες και δεξιότητες που θα μπορούσαν να προσφέρονται από τα σχολεία, όπως βλέπουμε σε άλλα κράτη, μπορούν να φέρουν καλά αποτελέσματα και να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των νέων. Η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών, η ελεύθερη κυκλοφορία των νέων, είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της ενιαίας αγοράς. Μπορεί να εξυπηρετήσει συμφεροντορισμένων πολυεθνικών, αλλά οπωσδήποτε εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί μπορούν έτσι να βρίσκουν καλύτερες θέσει εργασίας, ίσω και σε άλλες χώρες βεβαίως, εάν έχουν τις σχετικές δεξιότητες στην εκπαίδευση. Είμαι πεπισμένο λοιπόν, απολύτω πεπισμένο, ότι αυτές οι αποκλήσει, αυτά τα κενά που μερικέ φορέ αναδεικνύονται, οι διαφορές μεταξύ βόρειων, νότιων, ανατολικών, δυτικών κρατών θα καλυφθούν λόγω της διακίνησης των ανθρώπων, λόγω της κυκλοφορίας τους. Και εδώ έρχεται να υπηρετήσει το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη εκπαίδευση, προσφέροντάς του το καλύτερο δυνατό επίπεδο εκπαίδευσης σε, προσιτό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορεί να ξεπεράσει τα κοινωνικά εμπόδια ή χάσματα, προσφέροντας δηλαδή εκπαίδευση της κατάλληλης δεξιότητας και την ευκαιρία για κοινωνική κινητικότητα. Αυτή είναι η δουλειά μας πιστεύω. Και στηρίζομαι στη δική σας υποστήριξη για τη δραστηριότητα αυτή, ώστε να προσφέρουμε και καλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον στους νέους. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Στο δεύτερο γύρο. Επτά συναδέλφοι έχουν στήσει το λόγο. Παρακαλώ ο καθένα να περιοριστεί στα δύο του πολύ λεπτά. Και πιο σύντομα βεβαίω, αν θέλετε, καμία αντίρρηση. Και εσεί, κύριε Επίτροπε, αν θέλετε, όσο το δυνατόν πιο σύντομα τι απαντήσει σα, για να μπορούμε να ακούσουμε όλου του συναδέλφου. Κυρία Λιμπάτσικα, Κριστίνα. Ευχαριστώ. Επίτροπε, Άκουσα με μεγάλη προσοχή την παρουσίασή σας, τις ιδέες σας, τα οράματά σας για την εκπαίδευση. Υπάρχει κάτι που με ανησυχεί όμως. Δεν είπατε τίποτα για τους δασκάλους, για τους καθηγητές. Δεν είπατε ούτε μία φράση για την ομάδα αυτή εργαζομένων. Πώς σκοπεύετε να στηρίξετε τους δασκάλους και καθηγητές στην Ευρώπη για να προετοιμαστούν για το νέο ρόλο τους στο μέλλον πώς ερμηνεύεται τη σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ευχαριστώ. Σύντομες και συγκεκριμένες ερωτήσεις, σύντομες και συγκεκριμένες και οι απαντήσεις. Yes, it's my, it's my mistake. Ναι, λάθος μου ήταν. Η θέση των δασκάλων είναι πολύ σημαντική για την μελλοντική ανάπτυξη της ε, εκπαιδευτικής πολιτικής. Γι' αυτό έχουμε ειδικά ε, κονδύλια στο Εράσμους για την κατάρτιση των καθηγητών και μετακπαίδευση των καθηγητών, καθώς και την κινητικότητά τους. Και θα χρησιμοποιούσαμε τα εργαλεία, ηλεκτρονικά εργαλεία για να ενισχύσουμε την ε, ποιότητα της εκπαιδευτικής δασκαλίας και την κινητικότητα των δασκάλων. διασύνδεση του Ευρωπαϊκού Χώρου Πανεπιστημίων ή Ανωτέρων Σχολών, κύριε Λιμπάσκα. Έρευνα και ανώτερες σχολές, ναι. Well, the link is, uh, Η σχέση, ο σύνδεσμος είναι προφανής. Αν θέλουμε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, θα πρέπει να φτιάχνουμε προγράμματα, να έχουμε ομάδε για την κατάρτιση των δασκάλων και τη συνεργασία των δασκάλων. Και για τη δασκαλία των ευρωπαϊκών αξιών, των ευρωπαϊκών σπουδών, πληροφορίε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα πρέπει να συνδέσουμε τις, τις διάφορες κοινότητες καθηγητών που υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη μεταξύ τους, να τις δικτυώσουμε. Η κυρία Σόιντροβα. Θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω σε αυτό ρώτησε η κυρία Λιμπάτσκα. Δηλαδή συγκεκριμένα για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Κύριε Επίτροπε, το αναφέρατε ήδη και θα ήθελα να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα πώς το έχετε ε, σχεδιάσει αυτό, πώς μπορούν δηλαδή ορισμένα πανεπιστήμια να πάρουν ευρωπαϊκό χαρακτήρα. γιατί θεσπίζονται, πιστοποιούνται σε μια χώρα, παραδείγμα τα πανεπιστήμια. Με ποιο τρόπο θα πάρουν την πιστοποίηση ότι είναι ευρωπαϊκά. Πώς θα πάρουν το δικαίωμα να αναρτούν τον όρο ευρωπαϊκό. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ε, ιδιαίτερος ε, ευχαριστώ για την συνεργασία και τη δυνατότητα για εξασφάλιση ε, συνενετικά της ε, πρότασης αυτής. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το 29. Βεβαίως πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε. Είναι πολύ καλό πλέον να μην ε, εξαρτάται από την χρηματοδότηση του Erasmus Plus που αφορά την εκπαίδευση, αλλά να αποκοπεί από αυτό, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με την αλληλέγγυα και εθελοντική εργασία. Ερωτώ λοιπόν, μια και δεν αναφέρεται συγκεκριμένα το ποσοστό ε, κάλυψη σε σχέση με την εθελοντική εργασία από, και ποιο κομμάτι θα, πάει από το, θα χρηματοδοτηθεί από τις ε, ε, πιστώσεις που αφορούν ε, την επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη. έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση, γιατί αλλιώ υπάρχει κίνδυνος για, για τη σαφήνεια ποια προγράμματα θα μπορούν να χρηματοδοτούνται. Ευχαριστώ, Επίτροπο. Θα είμαι σύντομος. τα σχέδια για ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν δύο πυλώνες. Πρώτον, την ποιότητα. Γιατί θα πρέπει να διατηρήσουμε την ποιότητα και να μην την πλήξουμε στο βωμό της δημιουργίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Και ο άλλος πυλώνας είναι η συμμετοχικότητα. Δεν θα πρέπει δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε μόνο υπάρχοντα σχήματα συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων. Έχουμε δημιουργήσει δύο ομάδες εργασία. Η μία το, μεταξύ των εθνικών υπουργείων που είναι υπεύθυνα για την ανώτατη εκπαίδευση και η δεύτερη ομάδα εργασία ε, που απαρτίζεται από τους ε, έχοντες ε, συμφέρον για τους, από τους εμπλεκόμενους. Και εξετάζουμε αυτούς τους δύο πυλώνες, ποιότητα και συμμετοχικότητα. Θα είμαστε έτοιμοι το φθινόπωρο, γιατί οι πρώτες προσκλήσει εκδήλωση ενδιαφέροντος θα δημοσιευθούν τότε. Και το 2019 θα ξεκινήσουμε το πρώτο, την πρώτη πιλωτική φάση του προγράμματος Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Με τρία ως πέντε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σε αυτή την πρώτη πιλωτική φάση. Και στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 τα προγράμματα αυτά θα ε, λειτουργήσουν κανονικά πλέον. Θα δούμε στις αρχές του φθινοπόρου λοιπόν πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτών των προγραμμάτων. Τώρα για το Ευρωπαϊκό ε, Σώμα Αλληλεγγύης, ο προτινόμενος κανονισμός δεν προβλέπει διάκριση δραστηριοτήτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευελιξία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Στόχος μας 350.000 νέοι που θα, θα αυξήσουμε λοιπόν τις δραστηριότητες εθελοντισμού και υπέρ των δραστηριοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας και θα παρακολουθούμε ετησίως μέσω προγράμματος ε, ε, εργασίας ε, την εξέλιξη αυτού του προγράμματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε και εμένα μια ερώτηση για το σώμα αλληλεγγύης. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η πρόταση για το σώμα αλληλεγγύης θα στηριχθεί εν του 2021 στα όσα ήδη προβλέπονται ως προς το περιεχόμενο όμως, όχι ως προς την χρηματοδότηση, ως προς τους προσανατολισμούς. Γιατί δεν θα είχε νόημα βέβαια η συζήτηση, ο διάλογος που ολοκληρώσαμε με κόπο τώρα να πρέπει να ξανανοίξει του χρόνου. Ό,τι έχουμε καταφέρει μαζί μέχρι τώρα θα μπορούσε να παγιωθεί και να προχωρήσει ταχύτερα. Ίσως ακόμα και πριν τις εκλογές θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τον τριμερή διάλογο. Αν μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε, θα ήταν καταπληκτικό για να του δώσουμε σάρκα και ωστά. Άρα, από το νεύμα σας καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε. Παρακαλώ. Μια τα σχέδια της ε, Κομισιόν προβλέπουν αύξηση του προϋπολογισμού για τον αθλητισμό υπό το Erasmus Plus. Δεύτερον, επί δύο εβδομάδες ε, οργανώνω ένα πάνελ υψηλού επίπεδου για τον αθλητισμό. Θα ξέρετε την εκδήλωση αυτή, μιλάω για αυτήν, για να επικαιροποιήσουμε ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έχουμε ομοφωνία στο Συμβούλιο και προ το παρόν δεν υπάρχει. Ω εισηγητή για την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ολοκλήρωση της ε, σύμβαση. Ε, θα ήθελα να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο που υπάρχει σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Θα ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν ποια είναι τα επόμενα βήματα τη Κομισιόν, ούτω ώστε να βρούμε μία λύση για την κατάσταση αυτή. Τελευταία ερώτηση. Μία καλή λύση νομίζω ότι θα ήταν να έχουμε να γίνει μια επίσημη επίσκεψη τη Μάλτα, όλων των, ε, μιας αντιπροσωπείας μας δηλαδή, ε, και εσείς να συμμετάσχετε. Να πάει, λέει το Συμβούλιο, να επισκεφτεί τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Αθλητισμού της Μάλτας και να, τον, ε, να συζητήσει μαζί του για να υπάρξει λύση στο πρόβλημα. Θα ήταν ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα που θα έδινε το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να μπλοκάρει μια ολόκληρη διαδικασία για, για την προσπάθεια καταπολέμησης των στοιχημάτων, των στημένων παιχνιδιών, στον αθλητισμό κτλ. Ε, τι άποψη έχετε εσεί. Πώ μπορούμε να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο λόγω μάλτα. Ναι, πολύ σημαντική ερώτηση. Κύριε Επίτροπε. Ναι, θέλω να αυξήσουμε τον προπολογισμό για τα προγράμματα αθλητισμού. Επίση, ξέρετε πολύ καλά ότι προσωπικά είμαι πεπισμένο και προσπαθώ να ενισχύσουμε το προφίλ του αθλητισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τον αθλητισμό για όλους, πάνω απ' όλα. Γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χτίζει ομαδικό πνεύμα, κοινότητες, ενισχύει την αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορώ να πω Δεν μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένα ποσά. Θα ήθελα όμως ε, να αυξήσουμε αναλογικά τον προϋπολογισμό για τον αθλητισμό ε, στα πλαίσια του Εράσμους. Τώρα, για το, τα στημένα παιχνίδια. Θέλω να οργανώσουμε μία συμμαχία, όσοι επιθυμούμε να το καταπολεμήσουμε αυτό. Οι χώρες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι υπέρ της επικύρωσης να προσπαθήσουμε για να πιέσουμε την, ε, τις μαλτέζικες αρχές. Ήπια είναι αυτή η πίεση, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ. καλή αρχή θα ήταν όμως και να μπορούσαμε ίσως... Να μπορούσαν ίσως να ξεκινήσουν και οι 27. Παρακαλώ. Ναι. Ίσως θα μπορούσαμε να κερδίσουμε υποστήριξη για αυτά τα έργα και στα θέματα του πολιτισμού αλλά και του αθλητισμού εάν αναγνώριζαν το ενδιαφέρον της συμμετοχής σε αυτές τις δραστηριότητες, οι διάφοροι φορείς και περισσότερα χρήματα και η, επισήμανση των ε, εκδηλώσεων τους ως πολιτιστικών θα είχαν πολλά να κερδίσουν. Μπόσκο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο Στρασβούργο συζητήσαμε την, τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού συστήματος και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ότι οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στο διάλογο. Υιοθετήσαμε μάλιστα και μια έκθεση στην ε, οποία εντάξαμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, την Ευρωπαϊκή Διάση, Ευρωπαϊκές Αξίες, τη συμμετοχικότητα, τις οριζόντιες δεξιότητες. Νομίζω ότι ήταν πολύ θετική δουλειά που έγινε στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Και χαιρόμαστε που θα αυξηθεί κατά πολύ η χρηματοδότηση του Erasmus+. Ελπίζουμε ότι οι νέοι θα υποφεληθούν αυτών των νέων δυνατοτήτων που τους δίνονται. Συζητάμε εδώ και καιρό την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων σε θέματα γλωσσών, κοινέ εξετάσεις ε, γλωσσικών δεξιοτήτων κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε τα πράγματα σε αυτό το τομέα. Για παράδειγμα, μεγαλύτερη χρηματοδότηση για μαθήματα μηνωτικών γλωσσών, ε, λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την πολυμορφία της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ. Η πολυγλωσσία και η χρήση των γλωσσών από τις εθνοτικές μειονότητες είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πάντοτε πολύ προσεκτική στην προσέγγιση του θέματος αυτού. Κάποια στιγμή υπήρχε και ειδικό επίτροπος για την πολυγλωσία. Τώρα αυτό ο τομέας ανήκει στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, αλλά είναι κάπως υποτιμημένος. πρέπει μέσω του προγράμματος ε, Erasmus Plus ε, να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην πολυγλωσία. Θα θυμάστε ότι υπάρχει και μια πρωτοβουλία πολιτών η οποία θα φτάσει στην, θα εξεταστεί σύντομα νομίζω από την Κομισιόν αν επιβεβαιωθεί ο αριθμός των υπογραφών ε, η επίσημη διαδικασία θα οδηγήσει στην ε, έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας στο δεύτερο εξάμεινο του τρέχοντος έτους. Οπότε το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε σύντομα στην Κομισιόν. Στο ενδιάμεσο, προγράμματα του Εράσμους μπορούν να αυξήσουν χρηματοδοτικές δράσεις για την πολυγλωσία και την εκπαίδευση στην πολυγλωσία το σε ό,τι αφορά την αυτόματη αναγνώριση των διπλωμάτων, πανεπιστημιακών διπλωμάτων, ε, εκπαιδευτικών μονάδων κλπ. είναι μία από τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου. Θέλουμε να γίνει μια τέτοιου είδους αμοιβαία αναγνώριση, αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση. Έχουμε να προβλέψει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκών δεξιοτήτων και ένα πρόγραμμα μεταφοράς ε, εκπαιδευτικών μονάδων και αναγνώριση εκπαιδευτικών μονάδων, αλλά τελικά εξαρτάται από τα κράτη-μέλη το κατά πόσον θα εναρμονίσουν τα συστήματά τους και θα αναγνωρίζουν με αυτόν τον τρόπο αμοιβαία τα, ε, τις βεβαιώσεις και τα πτυχία. Στο τελευταίο Συμβούλιο Εκπαίδευσης τα κράτη-μέλη ε, ρητά υποστήριξαν την ιδέα της αυτόματης αναγνώρισης αυτών των ε, πτυχίων και βεβαιώσεων. Οπότε ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα υιοθετήσουμε ένα τέτοιο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Αλλά και από φοιτητέ του Εράσμους ε, μαθαίνουμε συχνά ότι η αναγνώριση των διαφορών σημείων ε, είναι βεβαίως προϋπόθεση για να μπορέσουν να μπουν στο ε, εξάμεινο του Εράσμου, αλλά ταυτόχρονα δεν αρκεί κιόλα και υπάρχουν πολλέ περιπτώσει όπου ε, τα πανεπιστήμια δεν αναγνωρίζουν τις, ε, τα πιστοποιητικά ή τα points που έχουν συλλέξει στο Πανεπιστήμιο Προελεύσεως τους οι φοιτητέ, όσο αξιέπαινα και είναι όσα έχουν γίνει, καταλαβαίνετε ότι και οι φοιτητέ αισθάνονται μεγάλη δυσφορία, γιατί αυτό το οποίο αποκομίζουν μετά από το εξάμεινο Εράσμου δεν αναγνωρίζεται στο οικείο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό σε ε, περισσότερα βήματα πρόοδου. Κύριο Σφέαρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητέ Επίτροπε, Στην αρχή της θητείας σας υπήρχαν πολλές αβεβαιότητες, Επίτροπε. Το πρόγραμμα άλλαξε άρδιν, υπήρξαν πάρα πολλές καινοτομίες, τα προγράμματα άλλαξαν άρδιν. Ε, και θέλω να σας συγχαρώ τελικά που ξεπεράσατε όλες αυτές τις δυσκολίες και μπορέσατε να φτιάξετε ένα πολύ καλό χαρτοφυλάκιο. Το Erasmus Plus λειτουργεί πάρα πολύ καλά πια και αξίζει περισσότερα κονδύλια. Έχετε διπλασιάσει την πρικοδότησή του. Η Επιτροπή Πολιτισμού θέλει περισσότερα λεφτά γιατί το ποσοστό απορρόφησης είναι πάρα πολύ καλό και η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από τα διαθέσιμα κονδύλια. Μία ερώτηση. Παρά το Brexit, μπορέσατε να αυξήσετε τον προϋπολογισμό φτάσατε σε συνένεση εντός της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό του προπολογισμού. Ποιο θα είναι το καθεστώ των φοιτητών στον Ηνωμένο Βασίλειο θα ήθελα να μάθω. Μιλάω για νέους, για τις οργανώσεις ε, και για όλους όσους θα επηρεαστούν από τον Brexit. Έχετε σκεφτεί το μοντέλο. Έχει υπάρξει κάποια συμφωνία. Δεν θέλω οι νέοι να βρεθούν σε χειρότερη θέση μετά τον Brexit. Μετά τον Brexit και θέλουν να υπάρξει μείωση της κινητικότητάς τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις ιδέες και λύσεις. Εξαρτάται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τη θέση του στις διαπραγματεύσεις. Μπορούμε να συζητήσουμε όλες τις εναλλακτικέ λύσεις και να βρούμε μια καλή λύση για εάν το Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνησή του δηλαδή, αποφασίσει τελικά. Τότε όταν αποφασίσει η κυβέρνηση του Βασιλείου για τον Brexit μπορούμε να το συζητήσουμε κι εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρουν και τι θέλουν, λέει η Πρόεδρος. Ο Λίτζιμ Μοργκάνο. Ευχαριστώ. Θα επικεντρωθώ σε ένα ερώτημα. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο Επίτροπος για τους φιλόδοξους στόχους και τα μέσα για να τους υλοποιήσουμε, που ήταν και το συμπερασμά του. Λαμβάνοντας υπόψη τώρα ότι μία από τις ευκαιρίες είναι μέσω του ορίζοντα 2020 και ειδικά για το ερευνητικό πρόγραμμα ε, το οποίο απασχολεί και ως εισηγητής για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού, νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή για να ανταλλάξουμε απόψεις, ε, για να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Έχουμε καταγράψει με θετικό πνεύμα ότι η Κομισιόν έχει προβλέψει ότι Χρειάζεται, μα χρειάζονται 100 δισεκατομμύρια για το νέο ε, πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στρατηγικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι υπάρχει υποεκτίμηση σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία. Αλλά ας ξεκινήσουμε αυτό το νούμερο, τα 100 δις. Η Κομισιόν δέχτηκε την πρόταση του Κοινοβουλίου και πρόβλεψε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε συνέργειες το είπατε και εσείς επίτροπε, μεταξύ ισχυών των προγραμμάτων και να συνδεθούμε, δηλαδή να συνδέσουμε το ορίζοντα και τα νέα προγράμματα, το νέο ε, πρόγραμμα Εράσμους, καθώς και το Δημιουργική Ευρώπη. Αυτά να τα συνδέσουμε. Αλλά διαπιστεύουμε με, διαπιστώνουμε με ανησυχία ότι ο πολιτισμός δεν θεωρείται πραγματική πολιτική προτεραιότητα ακόμα. Ε, γιατί έχει, είναι μειωμένη υποβαθμισμένη η θέση του, πέρα από τις προσπάθειες που κάνετε εσείς. Έτσι, πού θέλω να πω, ο συνολικό προπολογισμό για το δεύτερο πυλώνα, ε, συνολικέ προκλήσει τη κοινωνία, ανταγωνιστικότητα, βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, αυτό είναι ο τίτλο. Αυτό έχει αυξηθεί. Πολύ ωραία. Καλό είναι αυτό. Όμω υπάρχει και η προσέγγιση των πέντε κλάστερ δεν υπάρχει επαρκής, επαρκώς ισορροπημένη κατανομή των κονδυλίων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει, υπάρχει ένα κλάστερ ε, κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ασφαλής κοινωνία. Πέρα από το γεγονός ε, που μας ανησυχεί ότι προβλέπεται 2,8 δισεκατομμύρια, το ποσό αυτό δεν αρκεί για να καλύψουμε τις ανάγκες. Ε, και για να επανέλθουμε στην ψηφιοποίηση πολιτιστική κληρονομιά, διαφύλαξη της πολιτικής κληρονομιάς μέσω των νέων τεχνολογιών. Δεν φτάνουν αυτά τα 2,8 δις. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το μάτς που παίζουμε θα πρέπει να σε απασχολήσει περισσότερο. Η πρόεδρος με πιέζει με το χρόνο για την ανοιχτή ε, επιστήμη. Θα πρέπει να την χρηματοδοτήσουμε αρκετά. Μια στιγμή, πρόεδρε, να κλείσω υπάρχει το θέμα της μεγαλύτερης χρηματοδότησης για προγράμματα που αυξάνουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Παραδείγματος χάρη, έχουμε 100.000 ε, θαυμάσιους ερευνητές και αυτά είναι προγράμματα, ε, δηλαδή όπως το πρόγραμμα για την έρευνα, ας πούμε, που θα πρέπει να μας απασχολήσουν περισσότερο. Κάτι παραπάνω πρέπει να κάνουμε. Πάντα είμαι αυστηρή, γιατί είναι ζήτημα και δικαιοσύνης να μιλούμε ε, όλοι, να κάνουμε τις ερωτήσεις μας στο ίδιο χρονικό διάστημα για να έχουν όλη τη δυνατότητα να τις διατυπώσουν. Και αυτό είμαι και πιο αυστηρή στο θέμα του χρόνου. Έχετε το λόγο κύριε Πέτροπε. Ναι, συμφωνώ πολύ τόσο μαζί σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση και το σχέδιο θα προχωρήσει εφόσον βέβαια τα κράτη-μέλη είναι διτεθειμένα να διαθέσουν τα σχετικά κονδύλια. Αν μπορεί δηλαδή η Επιτροπή σας ή εσείς προσωπικά να πείσετε τα κράτη-μέλη να προσφέρουν περισσότερα χρήματα στα προγράμματα για τους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα προγράμματα για τους νέους της Ευρωπαϊκής πολύ ευχαριστώ να υποστηρίξω και μεγαλύτερη ακόμη ενίσχυση στο σχετικό προπολογισμό. Αλλά έχουμε τα διάφορα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στο το Marie Curie, Σροδόσκα που χρηματοδοτεί το χρηματοδοτούμε από τον ε, Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Το κέντρο, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, θα το είδατε ίσως ε, στην έκθεση που έγινε στο Μιλάνο, αν δεν κάνω λάθος, στη Ρώμη τα εξηγούσε όλα πολύ καλά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνεργασία, η σύνδεση των δραστηριοτήτων των ερευνητικών αυτών Ινστιτούτων και των πολιτιστικών ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θέλουμε βεβαίω και να αναπτύξουμε περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Κυρία Ροδρίκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Τρεις ερωτήσεις έχω. Πρώτα, μια πιο γενική. Πώς αντιμετωπίζετε γενικά τις περικοπές, ιδιαίτερα στη συνοχή και τη σχέση που υπάρχει, αν υπάρχει, ανάμεσα σε αυτήν την περικοπή και στην δυνατότητα αύξησης στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Πώς είναι δυνατόν η Κομισιόν να μην αντιλαμβάνεται ότι οι περιφερειακές ασυμμετρίες δημιουργούν και πολιτιστικές ασυμμετρίες. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, που είναι η μόνη χώρα του Νότου που βλέπει μειώσεις στη χρηματοδότηση, πολύ κακό όπως φαντάζεστε, γιατί έχουμε περάσει μια τρομακτική κρίση, αλλά ήθελα να σας πω, για αυτό που είπατε περί μείωσης της ανεργίας των νέων, πράγματι, από το 10,1 έχει πέσει το 7,9 ενέργεια των νέων στην Πορτογαλία. Όμως έχουμε δύο άκρους απομακρυσμένες περιοχές στην Ευρώπη. Ε, στην Μαδέρα 25% για ενέργεια των στις Αζόρες 24%. Αλλά και η Γαλλική Γουιάννα ε, είναι πολύ ανησυχητικό παράδειγμα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν θα ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας σε ό,τι αφορά το ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις άκρος απομακρυσμένες περιοχές, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα νέων ή καλλιτεχνών. Αν κάποιος θέλει να πάει από το Φουνσάλ της Μαδέιρα στην ε, Λισαβόνα, το ειστήριο κάνει 500 ευρώ ε, περίπου. Οπότε θα εφαρμόσουμε μια θετική διάκριση, όπως γίνεται και με, στα, και με τα όπως πρέπει να γίνει και για την έρευνα. 4 εκατομμύρια ευρώ για όλες τις άκρως απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης που έχουν μέχρι και 10 διαφορετικά πανεπιστήμια, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μικρό ποσό. Επίσης, θα πρέπει η επιμόρφωση των διδασκόντων να μην γίνεται αποκλειστικά με την τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία κάνει μεν θαύματα, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα, δεν είναι πανάκια. Yes, uh, the development, rural development. Η ανάπτυξη πέθρου και η ανάπτυξη των απομακρυσμένων περιοχών είναι μια από τις πιο σημαντικές μου ανησυχίες στην εκπαιδευτική πολιτική πράγματι. Υπάρχει μια έλλειψη στις υποδομές, στα σχολεία αλλά και στα πολιστικά ιδρύματα σε απομακρυσμένες περιοχές και σε περιοχές υπαίθρου. Ε, λείπει εξοπλισμός Υπάρχει μια υστέρηση λοιπόν σε ό,τι αφορά τι υποδομέ. Θέλουμε λοιπόν να συνδυάσουμε την πολιτική ανάπτυξη Πέθρου, ε, την περιφερειακή ανάπτυξη, ε, την πολιτική συνοχή και τα πολιτιστικά μα προγράμματα, έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά μα προγράμματα, έτσι ώστε πράγματι να ενισχύσουμε και τι υποδομέ αφενό, αλλά και να ενισχύσουμε επίση και την ελκυστικότητα αυτών των περιοχών στους νέους. Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε μια, ένα, ε, διαπραγματευόμαστε πιο συνολικά, πιο σφαιρικά εργαλεία που θα συμπεριλαμβάνουν όλα αυτά τα μία τα οποία σας είπα προηγουμένως, όλα αυτά τα εργαλεία που σας ανέφερα προηγουμένως, συνοχή, περιφερειακή ανάπτυξη, ανάπτυξη πέθρου κλπ. Έτσι ώστε η δράση μας να είναι πιο πλήρης, να μπορούμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό επιτόπου και ιδιαίτερα τους νέους. Σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση των διδασκόντων, των καθηγητών, ναι, αλλά θα δώσουμε έμφαση στην τεχνολογία. Γιατί η τεχνολογία εντάσσεται τόσο πολύ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, συζητούσα με μια Φινλανδή, η οποία μου είπε ότι είχε δύο παιδιά και μπορούσε να ε, ε, συγκρίνει το πορτογαλικό με το φιλανδικό σύστημα και οι διαφορές ξεκινούσαν ήδη από τις σχέσεις γονέων σχολείου, για να μην πάει πιο μακριά. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες διαφορές, ίσως όμως υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής σε ό,τι αφορά τις ε, μεθόδους επιμόρφωσης και θα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα τις ε, βέλτιστες πρακτικές που διαθέτουμε. Σα vielen, vielen herzlichen Dank, Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Επίτροπε για την καλή και εξαντλητική συζήτηση αυτής της τελευταίας ώρας, μια μισή ώρα περίπου. Ιδιαίτερα εγώ θέλω να τονίσω και να ξέρω το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα για το εράσμο σε κάθε γλώσσα. Πολύ ωραίο αυτό, εάν συμβαίνει. Αλλά ελπίζω με χρειαστεί και το επόμενο πρόγραμμα να περάσει πέντε χρόνια, χρόνια για να προσφέρει σε κάθε γλώσσα την δυνατότητα για συμμετοχή στο εράσμο. Η ασκούμενη που έχω εγώ έψαξε έκανε τον κόπο και έψαξε σε όλους αυτούς τους τομείς προγραμμάτων που μας ενδιαφέρουν εμάς ως Επιτροπή για να καταλήξει σε μια σειρά από ιστοτόπους που μεταφράζουν σε όλες τις γλώσσες μόνο τους τίτλους. Και όταν μετά έρχονται οι λεπτομέρειες πληροφορίες και τα σημεία είναι μόνο στα αγγλικά. Ε, αυτό ξέρουμε ότι είναι κοροϊδία. Διότι τα προγράμματα μας εδώ στην Επιτροπή μας είναι προγράμματα που απευθύνονται σε ανθρώπους και πρέπει οι άνθρωποι να είναι σε θέση να διατυπώσουν τις αιτήσει τους, αλλά για να τις διατυπώσουν τις αιτήσει τους πρέπει να είναι διαθέσιμες και στις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να απαιτήσω εγώ ένας μικρός αθλητικός σύλλογος για το τομέα του αθλητισμού στο Erasmus Plus να πρέπει να κάνει στα αγγλικά την αίτησή του για να εξασφαλίσει ένα 2.000 ευρώ Μπορεί. Στα ερευνητικά ε, Ινστιτούτα να θεωρείται αυτονόητο ότι μπορούν ή να απαιτείται κιόλας ότι θα μπορούν να μεταφράσουν ή να γράψουν στα αγγλικά μια αίτηση, αλλά μια μικρή πρωτοβουλία πολιτιστική, ένας αθλητικός όμιλος ε, μικρής ε, έκτασης. Αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν ως πολίτες στην Ευρώπη, που θέλουν να έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν και το ευρωπαϊκό ιδεώδες, την ευρωπαϊκή νοοτροπία τέλος πάντων, ε, δεν είναι δυνατόν να τους λέμε ότι θα είναι όλα στα αγγλικά. Τα έχουμε ετοιμάσει αν θέλετε, μπορούμε να σας τα δώσουμε γιατί τα έχουμε μελετήσει όλα και τα έχουμε έτοιμα αν θέλετε να τα δείτε σε ουσία στο τόπο όλα αυτά είναι εκτός από τους ε, υπερτίτλους στα αγγλικά. Αλλά σας παρακαλώ μεριμνήστε ώστε να είναι διαθέσιμα τα προγράμματα για τον πολίτη, για τον νέο, για τον πολιτισμό, να μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες, να έχει πρόσβαση ο πολίτης, να είναι προσβάσιμο. Ιδάλλως, αν δεν θέλει ο πολίτης, αν δεν είναι σε θέση τελικά να ε, αξιοποιήσει το πρόγραμμα, αν δεν είναι προσβάσιμο δηλαδή το πρόγραμμα, το πρόγραμμα στον πολίτη κατά τρόπο ευχερή, δεν χρειάζεται καν να συζητάμε για τα προγράμματα. Και πάνω απ' όλα, α μην περάσουν άλλα πέντε χρόνια για να είναι διαθέσιμα σε όλε τι γλώσσε. Κοιτάξτε λοιπόν, να το μελετήσετε, να το προσέξετε και να μεριμνήσετε πάντα και παντού να υπάρχουν όλες οι γλώσσες, οι 24 γλώσσες. Είναι απαραίτητο, είναι σημαντικό. με ό,τι φιλοδοξίες έχουμε ότι θα πρέπει στο μέλλον όλοι να μιλούν ε, τρεις γλώσσες λοιπά. Πολύ, ωραίος, πολύ ωραία η φιλοδοξία, αλλά πάντως στο άμεσο μέλλον δεν τη βλέπουμε να υλοποιείται. Επομένως πρέπει και αυτό να γίνει και σας καλούμε να το φροντίσετε και να κοιτάξετε πράγματι πού υπάρχουν τα προβλήματα, πού δεν λειτουργεί καλά αυτό το σύστημα. Για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες πιστεύω μπορούμε να έχουμε διάφορες συζητήσεις επιπλέον για τα επιμέρους ε, προγράμματα. Αύριο έχουμε, όπως είπα, και τις συζητήσεις με τις ε, υπηρεσίες για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, για το πρόγραμμα Εράσμους. Συζητήσεις θα γίνουν ε, βέβαια και με τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να αγωνιστούμε πιο σκληρά για τα διάφορα προγράμματα, να εξασφαλίσουμε περισσότερα κονδύλια. πιέζοντας και τα κράτη-μέλη για τα ποσά αυτά, γιατί είμαστε βέβαιοι ότι πρόκειται για χρήματα που υποστηρίζονται με ευρωπαϊκά χρήματα και προσφέρουν πραγματική προσθέμενη αξία. Και εδώ έχουμε να κάνουμε και με τριπλασιασμό, όπως είπαμε, ε, του ε, προϋπολογισμού της προκοδότησης για το Erasmus+. Είναι κάτι το οποίο δεν είμαστε τεθειμένοι να εγκαταλείψουμε ως στόχο και φαντάζομαι ότι αν καταφέρουμε να πείσουμε και τα κράτη-μέλη, η Επιτροπή δεν θα έχει καμιά αντίρρηση να διαθέσει περισσότερα κονδύλια για το μέλλον. Και αυτό ισχύει βέβαια όχι μόνο για το Erasmus Plus, αλλά και για το Δημιουργική Ευρώπη. Θα δούμε πόσο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Οι συγκεκριμένε συζητήσει θα συνεχιστούν. Σα ευχαριστώ και πάλι θερμά για την παρουσία σα σήμερα εδώ, για την πρωτοβουλία, για την προαγωγή ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. Αξίζει πραγματικά τον κόπο και οπωσδήποτε πρέπει να πείσουμε και τα κράτη-μέλη να μην αρχίσουν ε, να φωνασκούν ε, επικουρικότητα, τα χέρια κάτω από, το, ε, από την εκπαίδευση κτλ. Νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα αν συνεργαστούμε μαζί, περισσότερο μαζί και καλύτερα μαζί. Είναι σπουδαίος ο στόχος. Μπορούμε μαζί να τον υλοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρωτοβουλία λοιπόν. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία και ελπίζω πια τα κράτη-μέλη να αφήσουν τα ωραία λόγια και να προχωρήσουν και στις πράξεις. Ευχαριστώ πολύ. Και θα έρθει μέρα που θα τα ξαναπούμε, όπως λέμε. So, dann kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt. Και έτσι περνώ στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης για σήμερα. Σχέδιο γνωμοδότησης για τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάχιστα πρότυπα, γνωμοδότηση της Επιτροπής για την Επιτροπή Λίμπε, συγγνώμη, που έχει την αρμοδιότητα με την έκθεση πρωτοβουλία για τα ελάχιστα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τι μειονότητε. Εδώ Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε συμμετοχή με το άρθρο 54. Δεν τα καταφέραμε όμως. Δυστυχώς δεν ε, έγινε δυνατό αυτό. Παρόλα αυτά όμως η ΛΥΜΠΕ μας επέτρεψε μια στενή συνεργασία έστω και με τη γνωμοδότησή μας. Ο Ανδρέα Μπόσκορ έχει αναλάβει τη γνωμοδότηση αυτή, θα του δώσω τον λόγο. Έχει οριστεί η προθεσμία για τροπολογία για η προθεσμία για τις τροπολογίες 22 Ιουνίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας προβλέπεται για το Σεπτέμβριο. Κυρία Μπόσκορ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, και πέντε λεπτά το πολύ. Ναι. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που ε, επεξεργαζόμαστε αυτή τη γνωμοδότηση και θα μπορέσουμε έτσι να συνεισφέρουμε στο θέμα της, ε, της πολυγλωσσίας, της γλωσσικής ποικιλομορφίας. Ως ε, εισηγήτρια της ε, ΛΥΜΠΕ πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα θέματα των ε, μειονοτήτων, των προσφύγων, των ξένων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 50 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούν μια μειονοτική γλώσσα. Και σαν να τους κρύβουμε κάτω από το χαλί. Η έκθεση Αλφόνση το 2013 πραγματευόταν παρόμοια θέματα. Και πιο πριν, η προηγούμενη έκθεση χρονολογείται από το 2003. Άρα λοιπόν ήταν, είχε έρθει η ώρα να μιλήσουμε ξανά για τις μειονοτικές γλώσσες και τις περιφερειακές τοπικές γλώσσες. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να θέσουμε όλα τα θέματα που θέλαμε διότι το πεδίο Τη έκθεση έχει περιοριστεί, όμως θα υποβάλουμε τροπολογίε. για θέματα που δεν έχουμε συμπεριλάβει. Δεν υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση των ε, μειωνοτικών γλωσσών και των παραδοσιακών γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πολλούς αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. δεν υπάρχει καν κοινό ορισμό. Κάποιοι λένε ότι αυτό, ούτε αυτό είναι κακό. Όμως πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα κοινό ορισμό ε, προκειμένου να βοηθήσει αυτό το νομοθετικό μας έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία του Safety Pack, για παράδειγμα, έχει βοηθήσει. Στο δεύτερο σημείο της έκθεσης, κάνουμε λόγο για το, τη σύμβαση της, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και το Συμβούλιο της Ευρώπης ήδη έχει λοιπόν αυτή την σύμβαση πλαίσιο, αλλά και, άλλες, και άλλα κείμενα, των Ευρωπαϊκό Χάρτη Γλωσσών, Μειονοτικών Γλωσσών, συγγνώμη, ε, όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν βάση και να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. ζητούμε από τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν, να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν αυτά τα κείμενα του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Τα κριτήρια τη Κοπεχάγη, από την άλλη μεριά, εφαρμόζονται σε κράτη τα οποία επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπουν την προστασία των ε, εθνοτικών μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους, ιδιαίτερα των δικαιωμάτων τους. Οπότε, όμως τα παλιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρακολουθούν το σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων. Οπότε χρειάζεται ένας τέτοιος μηχανισμός και για τα παλαιότερα μέλη της Ένωσης. Ετησίως θα πρέπει να ε, υποβάλλονται ε, εκθέσεις σε ό,τι αφορά το σεβασμό των μειονοτικών γλωσσών σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μπορούμε να παρακολουθούμε από κοντά το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εκπαίδευση, Βέβαια, για παράδειγμα, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχει, ε, υπάρχουν ειδικοί κανόνες, νομοθετικά κείμενα. Ε, το θέμα είναι πάρα πολύ ευρύ. Για παράδειγμα, σε μειονοτικές γλώσσε, χρήση μειονοτικών γλωσσών στην διοίκηση επίσης ε, ή στις αθλητικές αναμεταδόσεις. στον τόπο τον οποίο διαμένουν οι μειονότητες ενδεχομένω, πινακίδες, ε, δίγλωσσες ε, ή έντυπα, διοικητικά έντυπα τα οποία θα είναι σε δύο γλώσσες κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδη. Παρακαλώ. Κυρία Ροντρίγκη, πρώτα. Μέχρι τρία λεπτά παρακαλώ. Τα Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητε άμεσα αρμοδιότητε για αυτά τα θέματα, Όμω η Χάρτα των ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ε, η έκθεση ε, όμως τύχει σημαντικά θέματα που αφορούν άτομα τα οποία ανήκουν σε τέτοιες μειονότητες στην, Ευρωπαϊ... στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες έτσι ώστε να ενταχθούν στις κοινότητές μας και γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να τηρούν τα οικονομικά πολιτιστικά κοινωνικά και γλωσσικά δικαιώματα των μειονοτήτων. Αλλά δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτό. Θα πρέπει να είμαστε πιο δραστήριοι, να προωθήσουμε τις κουλτούρες των μειονοτήτων, διότι αυτές ε, αποτελούν πλούτο για τις κοινωνίες μας. Η εκπαίδευση έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Η έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ήδη αναφέρεται στο δικαίωμα λήψη εκπαίδευσης ως απαραίτητο για την ανάπτυξη αυτών των μειονοτητών Νομίζουμε ότι η εκπαίδευση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτών των ατόμων. Ο ρόλος της εκπαίδευσης έχει άμεση σχέση με τη δράση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή οι αρχές οι οποίες βρίσκονται γεωγραφικά πιο κοντά στις μειονότητες είναι αυτές από τις οποίες θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να τους δώσουμε οικονομική και λειτουργική αυτονομία επαρκή έτσι ώστε να, πετύχει, πετύχουν το στόχο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία. Δεν θα πρέπει θα πρέπει να προασπίσουμε τα δικαιώματά τους χωρίς όμως να ε, υπερβάλλουμε δημιουργώντας ε, ε, ε, ψευδείς ελπίδες και καταστάσεις. Στις πολιτικές εκπαίδευσης για το θέμα του φύλου επίσης θα πρέπει να ακολουθούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το ότι ζητάει από την Κομισιόν να υποβάλει μια πρωτοβουλία για την ε, πολιτιστική πολυμορφία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ καλή πρόταση. Evans, bitte. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Τηρήστε και το χρόνο σας, κυρία Evans. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομη θα είμαι. Ευχαριστώ την εισηγήτρια πολύ καλές συστάσεις τη Μπορεί να ενταχθούν στην ε, έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Είναι σημαντικό ε, σημαντικά θέματα αυτά που είπατε και όσοι έχουμε ε, ασχοληθεί με αυτά τα θέματα ζητούσαμε αιτήσια παρακολούθηση. Ε, Αυτό το σημαντικό είναι, θέμα που έχει και για μένα σημασία, γιατί είμαι Ουαλή, 20% του πληθυσμού ε, χρησιμο... Ε, την Ουαλική γλώσσα, είμαι από δίγλωση κοινότητα και είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τη μητρική γλώσσα. Ε, εμείς Έχουμε μέτρα υποχρεωτικά για τους δημόσιους φορείς, ε, πρέπει να χρησιμοποιούν την, ε, τα ουελικά, αλλά αυτό δεν καλύπτει και τα, τις ιδιωτικές εταιρείε. Θα πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε άτομα που δεν μιλούν τις επίσημες γλώσσες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα ουαλικά και να τους διαφοροποιήσουμε με τις εθνικές μειονότητες, γιατί είναι τελείως διαφορετικό θέμα. Βεβαίως πρέπει να τα συμπεριλάβουμε και τα δύο, και τις δύο αυτές ομάδες. Επίσης ε, υπάρχει ένα ψηφιακό χάσμα. Θα το συζητήσουμε στην αυριανή μου έκθεση. Και θα ήθελα μία αναφορά στη συμπερίληψη των μειονοτήτων ε, στο Erasmus Plus και στο Δημιουργική Ευρώπη. Είναι πράγματα, θα τα, θα τα συζητήσουμε και αύριο επίσης. Καλωσορίζω την αναφορά στα ΜΜΕ που ξέρετε πολύ καλά τη σημαντική επίπτωσή τους. Ε, θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες ε, για αυτά τα θέματα που σας ανέφερα, αλλά γενικά θεωρώ ότι η έκθεση είναι πολύ καλή. Ευχαριστούμε. Στους επόμενους ομιλητές τώρα, η Julie Ward, δύο λεπτά το πολύ. Um, I just want... Για τη νοηματική, παρακαλώ, θέλω να ρωτήσω κάτι, νοηματική γλώσσα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν μπορούν όλοι να επικοινωνήσουν μέσω του λόγου και θα πρέπει η νοηματική γλώσσα να αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα. Θα πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να ενθαρρυνθεί ο κόσμος να μάθει τη γλώσσα αυτή, τη νοηματική, όταν τα μικρά παιδιά ε, μαθαίνουν λίγο την ε, νοηματική πολύ τα πρώτα τους χρόνια, ε, τους αρέσει πάρα πολύ, διασκεδάζουν πάρα πολύ, γιατί χρησιμοποιούν όλο τους το σώμα Εγώ ότι μιλάω και ήταν, θεώρησα πάντα στη ζωή μου ότι ήταν σημαντικό να μάθω κάτι τέτοιο. Όταν δουλεύεις με ανθρώπους που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον λόγο, είναι σημαντικό. Ε, να ξέρεις κάποια άλλα, να έχεις κάποια άλλα προσόντα, κάποιες άλλες δυνατότητε ε, να επικοινωνήσεις. Υπάρχουν και οι κοφάλαλοι. Ε, είναι η γλώσσα των κοφαλάλων. Αυτή πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Δεν ξέρω αν θα ενταχθεί στην έκθεση, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό σημείο και ήθελα να το θέσω. Σίλβια Κώστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε η συνάδελφος. Ε, είναι σημαντικό να δούμε και τις ε, γλωσσικές διαφορές ε, στην Ευρώπη. Ένα σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού μιλάει αυτές τις μειωτικές γλώσσες. Όπως είπε και η συγγήτρια, ε, χάρη στη Λισαβόνα, συνθήκη της Λισαβόνας, προχωρήσαμε. Γιατί η Λισαβόνα μιλάει και για τον γλωσσικό σεβασμό της και τις πιθανές παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών. Και μπορεί ε, να αποτελέσουν οι παραβιάσεις αυτές ε, βάση για να υπάρξει ε, παραπομπή της υπόθεσης επί παραβάση, με βάση το άρθρο 7. Συχνά λέμε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για να υπάρξει άμεση δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσει την ε, γλωσσική πυκλομορφία. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει το καθήκον αυτό από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ειδικά για αυτούς ε, που επικύρωσαν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις υπέρ αυτών των πολιτών. Επίσης, δύο πρωτοβουλίες των πολιτών δεν έγιναν δεκτές το 2013 για το θέμα αυτό. Κάποια από τα αιτήματα όμως τα οποία ανέφερε η συγγήτρια είναι πολύ σημαντικά. Το να λάβουμε υπόψη το θέμα αυτό στα διαφορετικά ταμεία. Δεν είναι άμεση ευθύνη, ναι, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το αναγνωρίζουμε, αλλά είναι άμεση ευθύνη των κρατών μελών να σεβαστούν αυτέ τι αρχέ που αναφέρει και η συνθήκη, καθώ και η σύμβαση του Στρασβούργου. Κατά την άποψή μου, το να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει για να γίνουν βήματα προ τα εμπρό, για να υποστηριχτούν οι δράσει των κρατών μελών, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το δικαίωμα, είναι πολύ σημαντικό. Και χάρη στα προγράμματα. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική και λογική και συνεπή θέση. Ευχαριστώ. Ρίχνω καμιά ματιά γύρω-γύρω. Είναι η Επιτροπή. Θέλει να λάβει το λόγο, μήπω. Όχι. Κυρία Στην εκπαίδευση των περιφερειακών γλωσσών ε, ενδιαφέρονται πάρα πολύ κάποια κράτη-μέλη στι εθνικέ του γλώσσε που είναι στοιχείο ενότητα. Στη Γαλλία, παραδείγματο χάρη, ε, έχουμε 24 περιφερειακέ γλώσσε ε, και Μητροπολιτικές και 24 στα υπερπόντια, συν 28 γλώσσες ε, Κανάκ της Νέας Καλλιδονίας. Φαντάζεστε την, το πρόβλημα και τις περιπλοκές. Επίσης ε, κάποιες άλλες ε, μιλούνται σήμερα, ενώ κάποιες άλλες δεν τις ξέρουν καθόλου οι νέοι, ας πούμε, οι οποίοι μιλάνε μόνο την επίσημη γλώσσα. Τα κράτη-μέλη επίσης δεν έχουν επικυρώσει όλα την Ευρωπαϊκή Χάρτα των Περιφερειακών και Μειωτικών Γλωσσών, όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Επομένως είναι σημαντικό αυτό το κείμενο να υπενθυμίσει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν ε, τις γλωσσικές χρήσεις. Και είναι κρίμα που το κείμενο λέει ότι είναι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ε, άμεσα αρμόδια για θέματα των, που αφορούν τις μειονοτικές γλώσσες. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις παρεμβάσεις. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Ναι, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν για τη δεσπόζουσα γλώσσα. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε ένα κράτος μέλος να ε, λάβει υπόψη τη γλώσσα σε πολύ πολύ μικρής σε 100 ατόμων ας πούμε. Δυστυχώς χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Ωραία, τώρα είναι εντάξει. Σίγουρα θα πρέπει να διακρίνουμε την κατάσταση σύμφωνα με το μέγεθος, ε, σε συνάρτηση μάλλον με το μέγεθος της μειονότητας. Τα κράτη-μέλη έχουν την αρμοδιότητα να κάνουν αυτή τη διάκριση και να αντιμετωπίσουμε διαφορετικό τρόπο την κάθε μειονότητα. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπε η κυρία Ροντρίγκε, δεν θα πρέπει να απομονώνονται οι μειονότητε. Θα πρέπει οι μειονοτικοί να γνωρίζουν, να μιλούν τη δεσπόζουσα γλώσσα, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να προστατεύσουμε και τις μειονοτικές γλώσσες, χωρίς να, τις, να απομονώνουμε τους ομιλητές τους από την υπόλοιπη χώρα. Επίση, πολύ σωστά, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι φορείς θα πρέπει να εμπλακούν. Το έχουμε αυτό ως παράδειγμα. Γίνεται ήδη. Όταν έχουμε μια μειονότητα, παράδειγμα, που μπορεί να ζει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, το Τυρόλο, τότε εκεί για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή μπορούμε να έχουμε ε, τα έγγραφα, δημόσια έγγραφα σε δύο γλώσσες ε, ε, ή τις πινακίδες να, είναι, τις κάνουμε δίγλωσσες κλπ. Πράγματι. Έτσι ώστε η, τοπική ή μειονοτική γλώσσα να είναι προσβάσιμη σε όλους. Οι γλώσσες πράγματι θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο νομικό καθεστώς. Α, η, νοηματική, συγγνώμη. Το κατά πόσο η νοηματική πρέπει να συμπεριληφθεί μεταξύ αυτών των γλωσσών. Η νοηματική δεν είναι μία γλώσσα. Κάθε χώρα ε, έχει τη δική της νοηματική γλώσσα. Αλλά θα μπορούσαμε να την συμπεριλάβουμε, να πούμε στα κράτη-μέλη ότι σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει και η ε, νοηματική γλώσσα να χαίρει παρομοίων ε, προνομίων, ας πούμε, ή παρόμοιες, ε, παρόμοιου καθεστώτος. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και σίγουρα δεν θέλουμε εμείς να αφαιρέσουμε εθνικές αρμοδιότητες. Βέβαια, μερικές φορές υπάρχουν και γίνονται και ακρότητες. Υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες δεν σέβονται τα μειονοτικά δικαιώματα, δεν θα αναφέρω ονόματα χωρών, αλλά βλέπουμε, αρέα και πού, παραβιάσεις των μειονοτικών δικαιωμάτων, ενώ η προστασία τους ήδη αποτελεί υποχρέωση για τις υποένταξη χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν. Τροπολογίες, είπαμε 22 Ιουνίου 10 το πρωί, το επενθυμίζω. Ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία στους συντάκτες. 24 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε Αυτά για σήμερα. Καλό σας βράδυ. Αύριο το πρωί στις 9 και ψηφίζουμε. Και ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος, και εμείς ευχαριστούμε. Όπως σας είχα υποσχεθεί, λέει η Πρόεδρος, τελειώνουμε και νωρίτερα.